Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε την κοινή μας αυτή συνεδρίαση. Σημείο πρώτο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση αυτής. Δεν ξέρω αν έχετε προτάσεις τροποποίησης, δεν βλέπω. Καμία εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώσει Προέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων δεν έχω, δεν ξέρω αν έχετε εσεί. Ε, τρίτο. Α, καλωσορίζω την κυρία Βίκη Φόρτ, Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερική Αγοράς και τα μέλη της Επιτροπής και τα μέλη της δική μας Επιτροπής προφανώς. Συνεδριάζουμε απόψε εδώ από κοινού για να ακούσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία για ορισμένα στοιχεία που αφορούν συμβάσεις ε, για παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ε, μελέτη αντικτύπου σχετική. Το πρώτο τμήμα είναι αυτό και το δεύτερο είναι κάτι που θα προεδρεύσει η κυρία Φόρτ, η οποία της δίνω μέσα στο λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, γιατί ε, παρακολουθούνται και ηλεκτρονικώς ε, τα δικά μας θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε μια κοινή συνεδρίαση για ένα από τα βασικά ε, θέματα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Το πρώτο τμήμα είναι κοινή μας αρμοδιότητα. Θα συμπροεδρεύσουμε. Ε, έχουμε πάρα πολύ καλά συνεργαστεί στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, οπότε υποθέτω ότι θα συνεχίσει αυτή η ε, συνεργασία. Το βασικό είναι οι συνάδελφοι που έχουν ε, εμπειρία για το θέμα αυτό από διάφορες επιτροπές να μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή e-meeting. Ε, ε, αν δεν... Ε, το, το, το, κώδικα QR μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση της εφαρμογής ή meeting. Εν πάση περιπτώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχετε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της συνεδρίασης. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Φόρντ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Τιρκ Μάιερ, που είναι τμήματάρχης ε, του δικαίου ε, των συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, να μας πει ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, για την κοινή αυτή ε, συνεδρίαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, το ότι είναι κοινή η συνεδρίαση. Πιστεύουμε ότι μόνο εποφελής θα είναι για το ε, θέμα που έχουμε να εξετάσουμε. Είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας. Έχουμε, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε προχωρήσει πολύ τις διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε με τη δική σας συνεργασία. Θα ήθελα καταρχάς για το ψηφιακό περιεχόμενο να πω ότι είναι το πρώτο παραδοτέο στο πλαίσιο της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς και της ε, στρατηγικής της. Έχει εντοπίσει σημαντικά εμπόδια για την ψηφιακή αγορά με έναν πολύ συνολικό ε, τρόπο. Ποια, ποιος είναι ο πολιτικός, ποια είναι η πολιτική και η οικονομική λογική πίσω από όλο αυτό. Γιατί εμείς τα ποσοστά ανάπτυξη τη ψηφιακή αγορά τα συγκρίναμε ε, και είδαμε ότι βρισκόμαστε πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ένα τρίτο μόνο των καταναλωτών αγοράζουν διασυνοριακά σε σχέση με αυτούς που αγοράζουν στη χώρα τους και ένα τρίτο των πολιτών πολλούν διασυνοριακά σε σχέση με αυτούς ε, που πολλούν ε, στην χώρα τους το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και η όχι τόσο καλή του κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που μας καθυστερεί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό θα θέλαμε να το αλλάξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο στόχους λοιπόν. Ο πρώτος στόχος είναι ότι θέλουμε να επιτύχουμε πιο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δεν, δεν θα πουλούν μόνο στη δική τους τη χώρα, αλλά σε ολόκληρη την ενιαία ψηφιακή αγορά και συνεπώς μπορούν να αυξήσουν την αγορά τους, να τη διευρύνουν ε, και να είναι πλέον ανταγωνιστική και σε σχέση με τους έξω ευρωπαϊκούς εταίρους τους. Ε, θέλουμε να έχουμε πολύ υψηλά ενωσιακά ε, κριτήρια και προδιαγραφές για τις ηλεκτρονικές αγοραπολισίες. Όταν προέβημε στην, στη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου, είδαμε την οικονομική κατάσταση το νομικό κομμάτι είδαμε ότι υπάρχει ελάχιστη νομοθεσία σε επίπεδο ένωσης, ε, σε επίπεδο κρατών μελών είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση, γιατί το κάθε κράτος μέλος ακολουθεί διαφορετικό δίκτυο, δίκαιο συμβάσεων. Ε, ε, κάποια, θεο κάποια κράτη-μέλη τις θεωρούν ε, ε ηλεκτρονικές αγοραπολισίες, κάποιες ε, καλύπτονται από τις υπηρεσίες. Τα πράγματα είναι διαφορετικά από το ένα κράτος μέλος το άλλο και είναι διαφορετική και η αποζημίωση σε περίπτωση προβλημάτων. Υπάρχει λοιπόν μια αναδυόμενη τάση ε, μεταξύ πολλών κρατών μελών. Ξέρουμε όμως ότι πολλά κρατημέρια ασχολούνται με αυτό το θέμα και τους απασχολεί. Θέλουν και νομοθετούν πλέον για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και βλέπουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία που υπάρχει ε, η, ε, είναι υπότεξεργασία αυτή τη στιγμή. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο που καλύπτουν. Είναι όλες όμως υποχρεωτικές. Γι' αυτό μας είπαν ε, εμπορικοί σύλλογοι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πριν καταλήξουμε σε 28 διαφορετικά σύνολα ε, ε, κανόνων ε, δεξιά και αριστερά και δεν μπορούμε πλέον να γίνει, κάνουμε τίποτε, δεν θα μπορεί κανείς να πουλήσει πια τα προϊόντα του στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα για τα προβλήματα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Το πρώτο ε, θέμα είναι, για παράδειγμα, ότι αυτοί οι νόμοι διαφορετικοί δημιουργούν κόστος για τους καταναλωτές. Η αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική 70 εκατομμύρια καταναλωτές έχουν χρησιμοποιήσει τις τέσσερις μόνο κύριες κατηγορίες ε, ε μουσική, αντιβάιρους, ε, παιχνίδια και cloud ε, και έχουν όλοι ε, αντιμετωπίσει προβλήματα. Ένα στου τρει αντιμετωπίζει προβλήματα με το ψηφιακό περιεχόμενο. Μπορεί να είναι διαφορετικά βέβαια τα προβλήματα, όμως ε, συχνά υπήρχαν προβλήματα συμβατότητας, όπως για παράδειγμα χαμηλότερη ποιότητα, δυναμία πρόσβασης, παραποιημένο περιεχόμενο κλπ. Και μόνο 10% αυτών των 70 εκατομμυρίων ε, ε, έχουν αποζημιωθεί και συνεπώς έχουμε προβλήματα και οικονομικής φύσεως. Ένα ακόμη θέμα το οποίο ε, έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ε, το ψηφιακό περιεχόμενο σε σχέση με τα δεδομένα που καλύπτονται ε, από αυτήν την, ε, ε, από αυτήν την πρόταση. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα βασικά επιτεύγματα της πρότασης αυτής. Το πρώτο πράγμα που εξετάσαμε βλέποντας την αγορά είναι ότι το ψηφιακό περιεχόμενο και τα δεδομένα που καλύπτονται είναι ένα τεράστιο μερίδιο της αγοράς, διάφορα σύνολα δεδομένων, αλλά αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι 30% έρχονται να αγοράσουν ε, ε, cloud ε, storage ε, ε, και 70% κάνουν streaming και πάνω από 50% βλέπουν ε, τηλεοπτικό περιεχόμενο και κατεβάζουν ταινίες. Πρόκειται λοιπόν για ένα τεράστιο μερίδιο αγοράς και καταναλωτές γνωρίζουν όλο και περισσότερο. Πάνω από το 80% των καταναλωτών γνωρίζουν ότι τα προσωρινά δεδομένα έχουν, τα προσωπικά δεδομένα έχουν μία οικονομική αξία, μια εμπορική αξία. Ε, δίνουν δηλαδή κάτι το οποίο ε, μεταφράζεται σε χρήμα. Πάνω από ένα στους τρεις, 36%, ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν πρέπει να παρέχουν κάποια προσωπικά δεδομένα και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο αυτοί οι καταναλωτές δεν μπορούν να έχουν τα ίδια ε, δικαιώματα με τους άλλους. Για παράδειγμα, ότι όταν κατεβάζει κάποιο κάτι που κάνει 0,99, ε, ένα τραγούδι για παράδειγμα, 0,99 ε, ευρώ, στο, στο παρελθόν αν κάποιο δηλαδή αγοράζει ε, χωρίς ε, ε, να, προσφέρει κάποια προσωπικά ε, δεδομένα, πρέπει να πληρώσει περισσότερο. Γιατί να συμβαίνει αυτό. Αυτό που θέλουμε εμεί να γίνει είναι να υπάρξει ένα ισότιμο ε, πεδίο ε, γιατί θέλουμε να αντέξει στο χρόνο η νομοθεσία μας το ψηφιακό περιεχόμενο και τα διάφορα μέσα παροχής του ε, είναι όλο και περισσότερο αόριστα και θέλουμε να υπάρξει ένας καλός σχεδιασμός των της διοχέτευσης του περιεχομένου αυτού, ώστε ε, να υπάρχει μια πιο ισότιμη κατάσταση και όχι πλεονεκτήματα για κάποιους και μειονεκτήματα για κάποιους άλλους. Αυτός λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές, ε, ο, αυτή είναι σε γενικές γραμμές η οικονομική και πολιτική μας λογική. Είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι μια στοχευμένη οδηγία πλήρους εναρμόνισης ε, μια οδηγία πλήρους εναρμόνισης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε τη δυνατότητα για ένα σύνολο κανόνων, βάσει των οποίων οι καταναλωτές μπορούν να πωλήσουν τα δεδομένα. Και επίσης είναι στοχευμένη, δηλαδή είναι μια προσέγγιση που ε, στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Είδαμε τα προβλήματα και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά και μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό η πρόταση ε, αφορά ε, ένα συγκεκριμένο ε, άρθρο ουσιαστικού ε, δικαίου που έχει 55 άρθρα ενώ οι άλλες υπηρεσίες καλύπτονται από νομοθετικό μέσο με 186 άρθρα. Θέλουμε λοιπόν να επικεντρωθούμε περισσότερο στα προβλήματα, όπως είπα, και προτείνουμε οδηγία και όχι κανονισμό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τους κανόνες αυτούς στα, στο δικό τους δίκαιο ε, συμβάσεων. Για παράδειγμα, δεν λέμε ποιο είναι το είδος της σύμβασης. Μπορεί τα κράτη-μέλη να πούν ότι είναι ε, ενοικίασης, ε, ε, υπηρεσιών. Δίνεται τέλος πάντων όμως η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διαλέξουν. Μπορούν να ενσωματώσουν αυτούς τους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία και συνεπώς δεν δημιουργείται πρόβλημα ε, με το εθνικό δίκαιο συμβάσεων. Πεδίο εφαρμογής. Πρώτη ομάδα εναρμόνισης αφορά μια ευ... έναν ευρύ ορισμό του ψηφιακού περιεχομένου Εξήγησα ότι θέλουμε να αντέξει στον χρόνο νομοθεσία, θα θέλαμε να είμαστε ουδέτεροι τεχνολογικά δεν θέλουμε διακρίσεις ανάλογα με την κατηγορία του ψηφιακού περιεχομένου ή τι δίωδο ε, μετάδοσής του ε, θα χρησιμοποιηθεί. Καλύπτουμε ψηφιακό περιεχόμενο σε ένα απτό μέσο, για παράδειγμα σε ένα CD, ένα DVD. Καλύπτουμε το λογισμικό που κατεβάζει κάποιος από το ίντερνετ, για παράδειγμα ένα πρόγραμμα Office. Καλύπτουμε επίσης ε, λογισμικό ε, streaming ή πρόσβαση στο ίντερνετ. Για παράδειγμα βλέπει κανείς ταινίες στο ίντερνετ ακούει μουσική στο ίντερνετ, ε, έρχεται, προσπαθεί να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ με κάποιο ε, τρόπο ή θέλει να αποθηκεύσει μέσω cloud ε, κάποια ε, πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια, κάποια, μια ευρύτερη κάλυψη ε, όσον αφορά το τι σημαίνει ψηφιακό περιεχόμενο. Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο έναντι δεδομένων, εξηγούμε τη λογική, αλλά είναι σημαντικό να λέμε ότι δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε ολόκληρο το ίντερνετ. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε κλικ στο Google ή στο YouTube ε, είμαστε ε, στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Το είδαμε από την πλευρά του μέσου καταναλωτή που δίνει δεδομένα και γνωρίζει όλο και περισσότερο ότι δίνει κάτι, ότι προσφέρει κάτι ξέρει ότι η διεύθυνση IP του ή τα δεδομένα του συλλέγονται και αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το ρυθμίζουμε αν κάποιος ας πούμε πρέπει να δει μια διαφήμιση για να έχει πρόσβαση σε ένα ιστότοπο. Και αυτό είναι κάτι που δεν το ρυθμίζουμε. Οπότε επικεντρωνόμαστε σε ορισμένα μόνο σημεία. Και επίσης ε, κάποια ε, δεδομένα που είναι απαραίτητα μόνο για τη λειτουργία της σύμβασης και όχι για δεδομένα τα οποία πρέπει να συλλεγούν επειδή υπάρχουν, ε, επειδή νομικά χρειάζεται ή επειδή πρέπει να παρέχει μια υπηρεσία. Για παράδειγμα, αν πάρει κανείς ένα χάρτη πλοήγηση, Προφανώ προφανώς πρέπει να ξέρει ο δορυφόρο που βρίσκεσαι διαφορετικά δεν μπορεί να σου πει από το σημείο α στο σημείο β πώς θα πας. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα είναι εκτό του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία ε, και αν ζητά κανεί μόνο αυτά τα δεδομένα δεν καλύπτεται από αυτήν την ε, οδηγία. Επίση, η δοκιμή συμβατότητα. Χρησιμοποιούμε μία εν μέρη νέα προσέγγιση. Δίνουμε προτεραιότητα σε υποκειμενικά ε, κριτήρια. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στη σύμβαση είναι αυτό που μετράει. Δεν θέλουμε να υπάρξει μία σύγκρουση μεταξύ των δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας ε, αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πηγαίνουν πίσω στον ε, κάτοχο των δικαιωμάτων, αλλά από τον νόμο μπορεί να δώσει κάτι το οποίο πηγαίνει πέρα από αυτό που μπορεί να παρέχει με, με κάποια σύμβαση. Οπότε προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση. Όμως έχουμε αναλύσει πολλές συμβάσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι είναι έτσι κάπως... Ε, ε, ε, σκοτεινές, κάπως αόριστες, ε, ασαφείς, γιατί δηλαδή λέει ότι αυτός που παρέχει την υπηρεσία ή το προϊόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας κλπ. κλπ. Επίσης δίνονται στον καταναλωτή κάποια δικαιώματα. Επιμένουμε στο επίπεδο της οδηγίας πολίσεων και κάνουμε κάποια προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος. Θα το πω αυτό ξανά στο τέλος της παρέμβασής μου. Να πω η επόμενη ομάδα ε, την οποία εναρμονίζουμε είναι πώς θα γίνεται η άσκηση αυτών των δεδομένων, ε, η μετατόπιση του άχθους ε, απόδειξης. Επίσης εισάγουμε κάποια άλλα δικαιώματα στην περίπτωση που για παράδειγμα ο καταναλωτής λαμβάνει ένα προϊόν και στη συνέχεια αλλάζει το προϊόν αυτό και μπορεί να ολοκληρώσει τη σύμβαση προκειμένου να διαλέξει κάποια άλλη υπηρεσία που είναι καλύτερη στην ίδια αγορά. Ε, επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να λύσουμε τα βασικά προβλήματα. Είναι περίπου 20 ε, άρθρα ουσιαστικού δικαίου Πρώτον, για να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο και να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ε, να έχουν πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη αγορά και συνεπώς να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Δεύτερον, περισσότερη εμπιστοσύνη για τους καταναλωτές γιατί ξέρουν ότι αν αγοράζουν σε μια άλλη χώρα έχουν ένα σύνολο δικαιωμάτων ε, και ένα ε, πολύ ψηλό επίπεδο προστασίας τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στανμάιερ. Τώρα θα ακούσουμε τους συνεισηγητές. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Φως, συνεισηγητή από την Επιτροπή Γιούρη. Άξελ, έχεις τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σταόντεν Μάιερ. Επί της ουσίας συμφωνώ με τους στόχους που περιγράψατε. Βρίσκω επίσης εξαιρετικό το γεγονό ότι μιλούμε για πλήρως, πλήρη ενερμόνιση γιατί στον τομέα των δεδομένων πολύ συχνά ξεπερνιούνται τα, τα όρια και τα σύνορα και θα έπρεπε να αποφευχθούν πάση θυσία τα διαφορετικά πρότυπα μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα ισορροπημένο δίκαιο μεταξύ των συμβαλόμενων μερών, αφενός δηλαδή να μην μειώσουμε την προστασία των καταναλωτών, από την άλλη όμως να μην τους δώσουμε και υπερβολικά πλεονεκτήματα. Θα πρέπει να το δούμε πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη αυτό. Ένα ερώτημα. Ε, όσον αφορά την ελευθερία σύναψης συμβάσεων, ε, πόσο, κατά πόσο θα είναι δεσμευτικά, δεσμευτικό το έργο μας ε, ή, αν θα πρέ, ή, ή μήπως τελικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και συζητήσεις ε, περί της σύναψης συμβάσεων και σε άλλους τομείς. Επίσης, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ε, προσαρμογή, με άλλες προτάσεις για την ενιαία αγορά, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και τα υλικά αγαθά. Ε, για την σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων. Υπάρχει, θέλω να πω, ανάγκη να υπάρχει συνέπεια και συνοχή. Πρέπει να το προσπαθήσουμε αυτό και ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια ε, εναρμόνιση. Επίσης, Αναρωτιέμαι αν ο όρος καταναλωτές ενδεχομένως είναι κάπως παραπλανητικός γιατί μιλούμε πάντοτε για ζητήματα που συζητίζονται με τις συμβάσεις και όταν μιλούμε για υπηρεσίες, πώληση, μίσθωση οι εθνικές νομοθεσίες δεν κάνουν, το λόγο, δεν κάνουν λόγο για καταναλωτές, αλλά για πολιτές και αγοραστές ή για παρόχους ή παραλήπτες υπηρεσιών. Ε, από αυτή την άποψη ε, δεν ξέρω κατά πόσο ο όρος καταναλωτές που χρησιμοποιείται είναι ο Επίσης, Συμφωνώ ότι θα πρέπει να, να ε, είναι η νομοθεσία μας ανθεκτική για το μέλλον. Για το άρθρο 2 όμως όσον αφορά τον ορισμό των, του ψηφιακού περιεχομένου υπάρχει διαφορά μεταξύ δεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες ε, παρέχεται και μια άλλη υπηρεσία. Μια, παρέχεται μια εργασία κατά, τον παραδοσιακό, κατά την παραδοσιακή έννοια που ενδεχομένως θα πρέπει να διακριθεί από την έννοια της, ε, των δεδομένων. Στο άρθρο 3 ε, μιλούμε μόνο για τις ε, σχέσεις B2C. Εγώ όμως αναρωτιέμαι πώς θα, πώς, πώς θα εμπίπτει σε αυτό το δίκαιο όμως κάποιος επαγγελματίας και πώς θα προκύπτουν αυτά τα νέα δικαιώματα στο 5.1 γίνεται λόγος για προσωπικά ή άλλα δεδομένα. Εδώ νομίζω ότι ενδέχεται να ε, προκύψουν προβλήματα όσον αφορά την, ε, τον βασικό κανονισμό για, τα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και τέλος, <clears throat> αντιστροφή της, ε, της υποχρέωσης απόδειξης στο, στην παράγραφο 3 ο καταναλωτής. Αν αποφασίσει να αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν, θα πρέπει ο ίδιος να, να φέρει την ευθύνη ε, για το ότι το προϊόν αυτό μπορεί να ενταχθεί στο δικό του τεχνολογικό περιβάλλον. Όμως αναρωτιέμαι, θα πρέπει ο ίδιος ο πάροχος να φροντίζει για κάτι τέτοιο ή ο καταναλωτής, ο παραλήπτης της υπηρεσίας. Οπότε νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει με κάποιον τρόπο να... δεν έχουμε πετύχει ακόμα την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του παρόχου και του καταναλωτή. Αυτά σε μια πρώτη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να ακούσουμε και την κυρία Κέπχαρτ ενδεχομένω. Ένα τρίλεπτο ή δυνατό παρακαλώ κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση αυτή, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τις ε, συζητήσεις που είχαμε την περασμένη θητεία. Μήπως να κλείνατε κανένα μικρόφωνο εκεί πάνω. Ευχαριστώ. Καλώς είναι σας. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν γίνεται να ακούμε δύο μιλητές ταυτόχρονα. Ε, ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι αυτό που είχαμε συζητήσει στην περασμένη θητεία το σεβάστηκε και πρότεινε αυτό το σύστημα και όχι εκείνο το εθελοντικό που δεν μας βοηθούσε ήταν ατελέσφορο, το κάνανε στην άκρη πια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ υψηλό επίπεδο της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλω να τα επαναλάβω όλα από την αρχή. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που πρέπει να ρωτήσω, ε, γιατί δεν τα έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται με το πεδίο εφαρμογής. Ε, γίνεται ένας διαχωρισμός από ε, το ψηφιακό περιεχόμενο και τα κινητά αντικείμενα. Τι είναι αυτό. Δεν μας πείθει πάρα πολύ. Ε, αυτή η έκθεση σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Αγιμό ε, προσφέρει μεγάλο πεδίο επικαλύψεων και πάρα πολλές φαιές ζώνες, όπου δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τώρα ποιο αντικείμενο ε, είναι επιγραμμικό εμπόριο και ποιο είναι εμπόριο συγκεκριμένων αντικειμένων. Γιατί έχουμε και το ίντερνετ πλέον των αντικειμένων, το Internet of Things, και δεν καταλαβαίνω πότε και πώς θα γίνει αυτή η διαφορά. Πώς θέλετε να το κάνετε. Παράδειγμα, το έξυπνο αυτοκίνητο που δεν λειτουργεί χωρίς λογισμικό, αλλά δεν είναι και λογισμικό γιατί είναι αυτοκίνητο. Ε, και τελικά τι είναι αυτό, πώς ορίζεται. Ε, τέτοια ζητήματα τίθενται. Ή ε, κάποια προϊόντα που προέρχονται από την τρισδιάστατη εκτύπωση. Είναι παροχή υπηρεσιών. Αυτό τι είναι, είναι αντικείμενο, επιγραμμικό εμπόριο. Ή ανήκει σε άλλη κατηγορία. Αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν και χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Ε, το δεύτερο, ε, κατά πόσο ε, είναι συμβατές ε, οι παροχές με το συμβόλαιο. Ποιε είναι οι συμβατικέ υποχρεώσει. Είναι κάτι που έχει ρητά συμφωνηθεί ε, στο Συμβόλαιο. Αυτό είναι προβληματικό γιατί κυμαίνονται τα πράγματα, υπάρχουν πολλέ διαφορέ. Και πού είναι ε, άρα η ε, πρόθεση, η σκέψη για την εναρμόνιση, αν διαφέρουν οι βασικέ προποθέσει και σε τέτοιο βαθμό για του καταναλωτέ άνδρε και γυναίκε υπάρχουν στοιχεία αντικειμενικά, όπως είναι το θεμητό συμφέρον και οι υπόλοιπε ε, προσδοκίες των ε, καταναλωτών δεν παίζουν ρόλο, που παίζουν ρόλο στις κανονικές συμβάσεις, στις υπόλοιπες εμπορικέ. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε και να τα ελέγξουμε. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο βαθμό εναρμόνισης. Κοιτάξτε, εγώ είμαι καταρχήν υπέρ της πλήρους εναρμόνισης, αλλά τελικά θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο και μόνο. Και άκουσα τον συνάδελφο Φως προηγουμένως που λέει ότι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, όπως την προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί. Ε, τότε να αμφισβητήσω και εγώ την πλήρη εναρμόνιση, άμα το πάει έτσι. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, πολύ συγκεκριμένα και όσο νωρίτερα τα λύσουμε και τα διευκρινίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο πιο γρήγορα θα δουλέψουμε. Σταματώ εδώ προς το παρόν γιατί βλέπω ότι έχει περισσότερο και έχω θέσει και αρκετά σημαντικά ερωτήματα που χρειάζονται απάντηση. So, in our Στις σημειώσεις μας αναφέρεται ότι η Κομισιόν θα απαντήσει στους συνσηγητές. Αλλά αν δεν έχετε αντίρρηση να ακούσουμε πρώτα τους βουλευτές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, πολλά μέλη των Επιτροπών μας που έχουν ζητήσει το λόγο. Ίσως θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να συλλέξουμε τις ερωτήσεις. Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Οπότε, θα πάμε σε ένα γύρο σκιωδών. Ο Ντέιβιτ Πάνοβερ έχει το λόγο. Δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ροζιέχ, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Πολλές είναι οι πρόοδοι εδώ, ιδιαίτερα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ε, Υπάρχει και ένα νομικό κενό ήδη γιατί λίγες είναι οι χώρες σήμερα που προστατεύουν τους καταναλωτές και στην ψηφιακή αγορά και το ψηφιακό περιεχόμενο. Ε, χαίρομαι για τις εφαρμογές που προτείνετε και συμπεριλαμβάνονται και συμβάσεις ε, και το αντάλλαγμα δεν είναι οικονομικό, αλλά, ούτε χρηματικό, αλλά προσωπικά δεδομένα. Χρειάζεται επαγρύπνηση, τα γνωρίζετε όλοι αυτά και γενική συνοχή ε, σε σχέση με το δίκαιο ε, και το δικαίωμα των καταναλωτών. Για να υπάρχει αντίστοιχη προστασία το επιγραμμικού με το μη επιγραμμικό εμπόριο. Τι έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι δεδομένη αυτή η συνέπεια και η συνέχεια. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα φυσικά με την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και υποχρεώσεις για το πώς χειρίζεται κανείς τα προσωπικά δεδομένα και πώς συνδέεται με το κείμενο το οποίο μας απασχολεί η εν λόγω οδηγία. Και μετά θα ήθελα να επιμείνω και σε κάποια άλλα σημεία που ε, χωράνε βελτίωση, ενίσχυση ιδιαίτερα η διαλειτουργικότητα. Αυτή η έννοια σήμερα στον ορισμό που μας δίνεται, πώς να το πω, εισάγει μια υποχρέωση συμβατότητας, όχι διαλειτουργικότητας. Για το πεδίο εφαρμογής χρειάζεται νομίζω και εδώ διευκρίνηση. Ε, όταν ε, το ψηφιακό περιεχόμενο είναι σε ένα φυσικό υπόστρωμα. Τι γίνεται, τι ισχύει και ποιο πεδίο εφαρμογής. Ε, χαίρομαι για την πρόταση να καλύπτει η οδηγία ως αντα... τις συμβάσεις που έχουν ως αντάλλαγμα ε, την παροχή προσωπικών δεδομένων θέλω να συμπεριφθούν και τα συμβόλαια όπου ε, συμπεριλαμβάνεται και μια παθητική ε, ανταλλαγή δεδομένων που τα δίνει ο καταναλωτής χωρίς να το καταλαβαίνει. Και για το κριτήριο συμβατότητας και τις προσδοκίες των καταναλωτών σήμερα μας παραπέμπεται στους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Υπάρχουν και άλλοι τομείς προστασίας των καταναλωτών και εκεί αυτό το στοιχείο των θεμητών ε, ε, προσδοκιών ε, του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους 1,5 λεπτό, παρακαλώ, να χρησιμοποιούν ε, από το χρόνο ε, για... Η κυρία Αν Βαν Πόισεντ είναι εδώ. Ναι, πράγματι, Βίκη, εκ μέρους του Ντάν, επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πιστεύει ότι οι καταναλωτές χρειάζονται ένα σαφές σύνολο δικαιωμάτων όταν ε, αγοράζουν ηλεκτρονικά εντό ευρωπαϊκή Ένωση Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια αγορά, ένα περιβάλλον στην αγορά αυτή που να βοηθά και τις επιχειρήσεις. Να υπάρχει το ίδιο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές όταν ε, αγοράζουν ε, ηλεκτρονικά ε, ή με συμβατικό τρόπο κάτι. η με συμβατικο τροπο κατι οι καταναλωτές ψηφιακού περιεχομένου πρέπει να καλύπτονται από τους ε, νόμους προστασίας των καταναλωτών σαν αγόραζαν απτά αγαθά ε, και να, ε, και να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων που θα καλυπτουθούν ξεχωριστά από μια ειδική οδηγία προστασίας δεδομένων. Υπάρχει επίσης το θέμα της ποσοτικοποίησης των δεδομένων. Ποιος θα το εξετάσει αυτό το θέμα, ε, αν μια χώρα μέλος αποφασίσει να μην νομοθετήσει. Ε, επίσης, ε, υποχρέωση διαγραφής περιεχομένου σε περίπτωση, ε, σε περίπτωση μη παροχής υπηρεσίας και το λέω αυτό κυρίως για υπηρεσίες όπως το TripAdvisor. Κύριο Ταμπάσκης δεν είναι εδώ, Άντωνη Σκόφες από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ώρες ε, ήμουν σε μία κρόαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της. Νομίζω ότι σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο και εμείς ε, είμαστε εμπλεκόμενοι φορείς ε, και Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμη και εδώ που χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προστασία. Πολύ σημαντικό είναι και καλό είναι να εστιαζόμαστε στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτό είναι ο ευρύτερο στόχο μα και πρέπει να το σκεφτόμαστε κάθε φορά που κάνουμε κάτι. Η εναρμόνιση τώρα των κανόνων των συμβατικών είναι βέβαια πολύ σημαντικό για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και προστασία και για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο ορισμός του ψηφιακού περιεχομένου και η συμπερίληψη ε, στοιχείων ε, παροχής περιεχομένου έναντι ε, μη χρηματικών αμοιβών ε, θα έπρεπε να ε, είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικοί οι κανόνες ε, όταν κάποιος ε, λαμβάνει μια υπηρεσία έναντι παροχή δεδομένων ή έναντι χρηματική αμοιβή. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που αγοράζουν ηλεκτρονικώς. Δεν πρέπει όμως και να γίνεται υπερβολική ρύθμιση. Πρέπει να υπάρχουν καινοτομίες. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Δεν, δεν υπερβήκατε το χρόνο σας. Ο κύριος Καβαντά. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ ε, κυρία και κύριε Πρόεδρε. Ε, καλοσύνη σας που μου δίνετε το λόγο χωρίς να το ζητήσω. Ε, δεν θα μιλήσω 1,5 λεπτό. Τρει ώρε περάσαμε με του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαφόρων ενώσεων για να βρούμε τι διάφορε ισορροπίε. Θέλω να πω το εξή. Το Κοινοβούλιο θα φροντίσει αυστηρά να είναι ισόρροπο το κείμενο υπέρ των ε, καταναλωτών που είναι συμβαλόμενα μέρη. Δεν ε, καταναλώνουν απλώς μια υπηρεσία. Δεύτερον, θα προσέχουμε πάρα πολύ την προστασία των προσωπικών δεδομένων γιατί έγινε κατάφορη και σαφής κατάχρηση από πολλούς παρόχους. Και ένα τρίτο που θέλω να πω βεβαίως θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ε, πώς ε, μπορεί κανείς να καταγγείλει κάποια σύμβαση μακράς διάρκειας. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά για ένα κείμενο που μας έφερε που φτάνει στην σωστή ισορροπία. 54 δεύτερα πρώτα δεν την επιτυχάνει αλλά την πλησιάζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος μιλητής είναι η κυρία Ντενή Ντεγιόγκ. Κύριος Ντεγιόγκ. Απουσιάζει. Ο κύριος Μαστάλκα. Απουσιάζει. Um, Ευχαριστώ. Οι πράσινοι πιστεύουμε και εμείς ότι είναι ε, πολύ καλή αυτή η πρόταση και έρχεται στο σωστό χρόνο. Πρώτον, ε, για την ε, διάκριση μεταξύ των δύο προτάσεων. Έχω smartphone, φαντάζομαι και εσείς. Και το ερώτημα μου είναι, πρόκειται για ψηφιακό περιεχόμενο σε υλικό μέσο ή υλικό αγαθό. Ή το ένα ή το άλλο. Αλλά είτε το ένα είτε το άλλο έχουμε πρόβλημα. Διότι με ένα, ένα κουμπί είναι πολύ σύνηθες να σπάσεις ένα smartphone. Εδώ έχουμε να κάνουμε με υλικό αγαθό. από την άλλη πλευρά, αν έχεις ένα smartphone που από άποψη υλικού εξοπλισμού λειτουργεί άψογα, αλλά έχει πρόβλημα το λογισμικό του, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Άρα ε, εγώ δεν θα έλεγα ότι λέει η αιτιολογική έκθεση, ότι το λογισμικό δηλαδή ε, ε, υπόκειται σε κάποιον. Μήπως θα έπρεπε το λογισμικό στο smartphone να εμπίπτει στην, ψηφιακή, στην πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο και το, ο υλικός εξοπλισμός του, του κινητού αυτού στην, στην άλλη πρόταση για τα υλικά αγαθά. Επίσης, ε, υιοθετούμε μια περίεργη στάση όσον αφορά τις υπηρεσίες. Ε, αλλά ε, για κάποιους, ε, κάποιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση στο cloud, ε, είναι υπηρεσίες. Μήπως όμως αυτό θα οδηγήσει κάποια κράτη-μέλη να ρυθμίσουν όλα αυτά τα ζητήματα ως υπηρεσίες ε, μήπως θα έπρεπε να, να υπάρχει ένα πιο, μια πιο ευρεία προσέγγιση για όλο το ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτά προς το παρόν περιμένω την απάντηση της Κομισιόν. Ο κύριος Μάρκο Τζούλο, όχι δεν είναι εδώ, είναι. Α, συγγνώμη. Δεν σας βλέπω, με τυφλώνει ο ήλιος. Ε, κύριε Τσούλο. Ε, ringrazio, ma passo. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα μιλήσω. Ε, ε, Η κυρία Φεράρα δεν είναι παρούσα. Τότε να πάμε στα άλλα μέλη των επιτροπών μας που έχουν ζητήσει το λόγο. Κάλλας, Ραπίνη, εγώ, Κάποιος άλλος που θέλει να μπει στον κατάλογο μιλητών. αέρα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα μόνο ζήτημα για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Και το ζήτημα αυτό αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Ε, όταν λύγει μια σύμβαση, ο καταναλωτής θα μπορεί να πάρει πίσω το ψηφιακό του περιεχόμενο. Εγώ συμμερίζομαι αυτόν τον στόχο τη επιτροπή, Αλλά η διατύπωση είναι ασαφή, γιατί μιλά ταυτόχρονα για ψηφιακό περιεχόμενο, δηλαδή μιλάμε για περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει ο ίδιο ο χρήστη, αλλά μιλά και για προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα. Εγώ νομίζω ότι οι καταναλωτέ χρειάζονται, φυσικά, ε, αν έχουν ανεβάσει φωτογραφίε να τι πάρουν πίσω, αλλά δεν χρειάζεται να πάρουν πίσω τα δεδομένα για το Πόσε φορέ ή σε ποιο level φτάσαν σε κάποιο παιχνίδι που είχαν καταβάσει σε εφαρμογή στο κινητό του. Όσον αφορά το δίκαιο για την προστασία των δεδομένων, οι εταιρείε θα πρέπει να ανωνυμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα. Αν ε, δεν ε, ε, ξεκαθαρίσουμε τι είδους δεδομένα θα παίρνουν πίσω οι χρήστες και τι είδους δεδομένα θα πρέπει να ανωνυμοποιηθούν, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Τι πιστεύει λοιπόν η Κομισιόν για αυτό το θέμα. Και κάτι για τις πλατφόρμες. Και το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες έχουν κάποια προσωπικά δεδομένα και κάποιες άλλες ε, πλατφόρμες έχουν για παράδειγμα δεδομένα πληρωμών αυτό το ζήτημα ε, πώς ακριβώς το χειρίζεται η πρόταση οδηγίας. Κύριε Γραπίνη. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σκέφτηκε να υποβάλει την πρόταση αυτή. Όπως είδαμε και από τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων, Πιστεύω και εγώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάποιους όρους ε, στο πλαίσιο αυτής της πρότασης ε, οδηγίας, το πεδίο εφαρμογή, όπως είπε και η Εύελιν. Ακόμη και αν πρόκειται για οδηγία και όχι για κανονισμό, χρειαζόμαστε κανόνες πολύ καλά καθορισμένους, ίδιους για όλα τα κράτη-μέλη, ακόμη και αν ε, γίνεται μετά μεταγραφή της νομοθεσίας ε, στην εθνική νομοθεσία των κρατών ε, μελών δεν θα καταλήξουμε σε τίποτε αν είναι διαφορετικοί οι ορισμοί που θα ισχύουν στα πολιτήρια συμβόλαια των 28 κρατών μελών. Θέλουμε να έχουμε εναρμονισμένους κανόνους, ε, κανόνες ενιαίους ε, και για τις πωλήσει στο διαδίκτυο αλλά και στις ε, κανονικές παραδοσιακές πωλήσει. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν είναι σαφή ακόμη. Thank you. I've got some very... Ευχαριστώ έχω και εγώ κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στο 3.1, τι εννοείται any other data. Τι ακριβώς εννοείται, τι, τι, τι εννοείται οποιαδήποτε άλλα δεδομένα. Στα, στο 5.2 μιλάτε για την παροχή περιεχομένου αμέσως. Αυτό όμως δεν είναι στον έλεγχο του ανθρώπου που κάνει την παροχή. Μπορεί να έχει να κάνει με την ε, σύνδεση του ίντερνετ, για παράδειγμα. Στο άρθρο 6 μιλάτε για περιεχόμενο που πρέπει να έχει ε, μια ποιότητα και μια ποσότητα που να διαρκεί ε, στο χρόνο. Τι ακριβώς εννοείται υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου για αυτούς τους όρους. έχει ε, γίνει εδώ πέρα μια αντιγραφή και επικόλυση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Έχετε στο μυαλό σας τα απτά ε, αγαθά και προσπαθείτε να μεταφέρετε τους ορισμούς στο ψηφιακό περιεχόμενο. Όσον αφορά τώρα την επιστροφή δεδομένων ε, από τους παρόχους, από το πρώτο κλικ πρέπει να γίνεται αυτό. Τι εννοείται δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της σύμβασης από τους ίδιους καταναλωτές. Τι θα πει αυτό, εννοείται δηλαδή δεδομένα τα οποία μπορεί να έχουν παραχθεί από το ε, κώδικα της πηγής, ότι πρέπει κάποιος για παράδειγμα να ε, εκχωρήσει κάποιους κώδικες του ήδη από πριν, εδώ θα έχουμε κάποια προβλήματα συμβατότητας τότε. Ε, δηλαδή πρέπει να γίνεται ανείχνευση του κάθε byte και του κάθε κλικ, γιατί αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους παρόχους. Και το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνδέεται όλο αυτό με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων και το CRD. I would also have a short question. Και εγώ έχω μια σύντομη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπάρχει νομολογία στο παρελθόν για αυτή τη διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των αγαθών ε, σε διασυνοριακές ε, ε, περιπτώσεις. Θα ήθελα να λάβει υπόψη της την ομολογία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να τη βοηθήσει όταν, γίνει, όταν θέλουμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ αυτών των δύο τομέων. Αν κατάλαβα καλά αυτό είναι το τέλος των ερωτήσεων, οπότε να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει. Ευχαριστώ. Μεγάλος ο κατάλογος. Θα προσπαθήσω να καλύψω όλα τα ερωτήματα. Αν ξεχάσω κάτι, ε, είμαι βεβαίω στη διάθεσή σας. Θα ξεκινήσουμε με τα ερωτήματα που ανέφεραν πολλοί ευρωβουλευτές, γιατί πρόκειται προφανώς για πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, υπήρξε ερώτημα για, το... για τη σχέση μεταξύ online και offline ε, πωλήσεων. Ποια είναι η σχέση ε, των προτάσεων μας ε, με τον κανονισμό για την προστασία των καταναλωτών και με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και γενικά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρώτον, η σχέση με την πρόταση για τις εξαποστάσεις και τις ηλεκτρονικές πωλήσει. Διαπιστώσαμε στην διαβούλευση, στη δημόσια διαβούλευση που έγινε πέρσι, ότι ε, ένα, ε, μία, μία από τις απαντήσεις ήταν ότι αν ε, ρυθμίσετε το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να ευθυγραμμίζετε η πρότασή σας αυτή με, το, ε, με την, οδηγία για τις πωλήσει προς καταναλωτές ε, αυτά βεβαίως και την πήραμε υπόψη εκτός από τις περιπτώσεις που είναι πολύ ιδιαίτερες ε, ε, και αφορούν μόνο το ψηφιακό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μιλάμε για τα 11 μέσα. Ε, υπάρχει η ίδια ιεράρχηση με την ε, οδηγία ε, για τις πωλήσει, αλλά υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά την επισκευή και την αντικατάσταση, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα στο ψηφιακό περιεχόμενο, γιατί στο ψηφιακό περιεχόμενο απλά θα πάρεις εκ νέου, θα πάρεις από την αρχή ένα καινούριο προϊόν. Δηλαδή προσαρμόσαμε την πρότασή μας στις ιδιαιτερότητες της του ψηφιακού περιεχομένου. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση τη πρότασή μα με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θεωρούμε ότι και οι δύο πράξει θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, και ε, θεωρούμε ότι, θα, ε, ότι καλύπτουν δύο διαφορετικές σκοπιές. Ο, η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πηγάζει από την προστασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών ελευθεριών, των ατομικών δικαιωμάτων, ενώ αυτή η πρόταση προσπαθεί να, να επιτύχει μία ε, ισορροπία κατά τη σύναψη συμβάσεων. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αν το προϊόν δεν είναι τόσο καλό όσο είχε υποσχεθεί ο πολιτής, θα πρέπει να έχω συγκεκριμένα ένδικα μέσα ή ε, ένα επίπεδο αποζημίωσης. καλύπτουν δηλαδή οι δύο προτάσεις μας διαφορετικά πράγματα, αλλά θα πρέπει να συνεπάρχουν. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε επίσης ότι και οι δύο πράξεις θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν αλλά χωρίς αυτό να δημιουργεί ε, επιπλέον βάρος στον πάροχο. Και βασική μας επιδίωξη είναι η εξής, ότι όταν έχουν δοθεί προσωπικά δεδομένα, η πρότασή μας λέει ότι ο πάροχος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα. Χρησιμοποιήθηκε αυτή η διατύπωση γιατί δεν καλύπτουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο είδος δεδομένων, πρώτον, και δεύτερον, ε, εξασφαλίζουμε μέσω τη λογική σκέψης ότι αν ο πάροχος έχει κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνει σύμφωνα με την, ε, με την οδηγία για, την προσωπική, για τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή να νομοποιήσει και να διαγράψει τα δεδομένα, τότε ε, ε, έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και τέλος, Όσον αφορά το, το ζήτημα της συνοχής ε, με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχει ε, συνέπεια διότι και οι, και δύο πράξεις αλληλοσυμπληρώνονται. Η CRD εναρμονίζει τις προσυμβατικές υποχρεώσεις ενημέρωσης και ε, τις, ε, τις ίδιες τις και καλύπτει όλα, όλες τις ε, συμβάσεις και κατά συνέπεια καλύπτει και όλες τις συμβάσεις που, συνάπτονται και εμπίπτουν εντός αυτής της πρότασης. Ε, εκτός από τις ε, συμβάσεις που συνάπτονται με αντίτιμο την παροχή προσωπικών δεδομένων. Εδώ μπορεί και να αναθεωρήσουμε την CRD. Δεν θέλαμε να αναθεωρήσουμε την CRD όταν κάναμε αυτή την πρόταση, γιατί η CRD ε, ε, ψηφίστηκε το 2011 και τέθηκε σε ισχύ το 2014. Είναι πολύ καινούργια ακόμα. Θα κάνουμε λοιπόν μια διαδικασία αναθεώρησης το 2016, αλλά θα ε, ε, εξετάσουμε ολόκληρο, όλες τις εμπειρίες ε, και σε αυτήν την πρόταση που σας παρουσιάζουμε εδώ θα, θα, θα ρυθμίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα που σας ανέφερα. Και ένα δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται με τον ορισμό του ψηφιακού περιεχομένου. Η CRD είναι κάπως διαφορετική γιατί περιορίζεται στις, ε, στις παραδοσιακές εμπορικές συναλλαγές. Αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν μόνο τρεις πολύ μικρές ε, διαφορές. Ε, όσον αφορά τις, τις προσυμβατικές υποχρεώσεις ε, ε, ενημέρωσης. Πρόκειται για πολύ μικρά σημεία που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης της CRD όταν έρθει ο καιρός. Για το δεύτερο σύνολο δεδομένων που έχουν ανακύψει, πώς θα αντέξει στο χρόνο αυτή η νομοθεσία ή τι ακριβώς εφαρμόζουμε. Κάτι που αναφέρθηκε ήδη από πολλούς βουλευτέ είναι το ενσωματωμένο λογισμικό. Η κυρία Γκέπχαρτ ε, αναφέρθηκε στο έξυπνο αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Ένα πλυντήριο για παράδειγμα. Ε, το, τα πλυντήρια σήμερα πια ε, λειτουργούν με λογισμικό. είχαμε τρει επιλε, ε, επιλογές. Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε του κανόνε για το ψηφιακό περιεχόμενο, για τι ηλεκτρονικέ και εξαρτάσει πωλήσει ή ένα μείγμα αυτών των δύο βασικά εμείς δεν θέλαμε να προχωρήσουμε σε ένα μείγμα των ε, δύο συνόλων κανόνων γιατί ε, προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση του μέσου καταναλωτή και το να έχεις μια ε, ανάμιξη των κανόνων μπορεί να είναι σαφές σε έναν δικηγόρο ή σε έναν νομικό αλλά άντε να εξηγήσει τώρα ότι σε έναν καταναλωτή ότι έχει διαφορετικά δικαιώματα δικαιώματα ανάλογα με το αν δεν λειτουργεί ο κάδος του πλυντηρίου του ή το λογισμικό του πλυντηρίου του. Εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής λύση και έτσι καταλήξαμε στην εξή λύση. Ε, έχουμε είτε τα υλικά ε, ε, αγαθά είτε το ψηφιακό περιεχόμενο. Και αυτό που θεωρήσαμε εμείς ότι θα αντέξει στο μέλλον είναι το εξή. Θα να βάλουμε δύο προποθέσει. Πρώτον, το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του αγαθού. Δηλαδή, σε ένα πλυντήριο το λογισμικό του αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πλυντηρίου. Και δεύτερον, αν η λειτουργικότητα του ε, ε, του ψηφιακού περιεχομένου υπόκειται στην ε, γενική λειτουργικότητα του αγαθού. Με άλλα λόγια, το πλυντήριο έπινε τα ρούχα μου. Να έρθω και στο παράδειγμα του αυτοκιν του αυτοκινήτου. Εγώ πριν από μερικού μήνε για πρώτη φορά μπήκα σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τόσο πολύ λογισμικό σε, αυτοκίνητο. Αλλά και πάλι το λογισμικό αυτό στόχο έχει να με, να με πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Ίσως στο μέλλον σκοπός του αυτοκινήτου ε, θα, θα είναι να είναι ένα γραφείο ε, πάνω σε τροχού ή ένα χώρο αναψυχή Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, αλλά θεωρούμε παρόλα αυτά ότι η πρότασή μας αντέχει στο μέλλον και νομίζουμε ότι η διάκριση που κάνουμε σήμερα ε, που ισχύουν οι κανόνες για, για τα αγαθά, σε 15 χρόνια μπορεί βεβαίως να καταλήξουμε σε ένα, σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Ότι μπορεί τέλος πάντων να υπερισχύουν οι κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο. Αλλά σήμερα από την σκοπιά του, του μέσου καταναλωτή θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες για τα υλικά αγαθά. Και δεύτερο στοιχείο που αναφέρθηκε από πολλούς ευρωβουλευτές είναι ότι το ψηφιακό περιεχόμενο βρίσκεται σε υλικό αγαθό. Δηλαδή το, η μουσική στο CD ή η ταινία στο DVD. Τι θα ισχύει. Και εδώ είχαμε τρεις επιλογές. Θα μπορούσαμε είτε να πούμε ότι υπάρχουν οι κανόνες για τα αγαθά ή υπάρχουν οι κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο ή μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση. Η διάκριση και εδώ θα ήταν η νομικά πιο σαφής ε, επιλογή. Αλλά για τους ίδιους λόγους δεν το κάναμε. Ε, ήταν στα πρώτα μας προσχέδια κειμένου ε, η επιλογή που είχαμε διαλέξει. Αλλά δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα αυτό το πράγμα στον μέσο καταναλωτή. Ε, γιατί θέλει να ξέρει, θα ισχύουν οι κανόνες για τα υλικά αγαθά ή οι κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και εδώ κοιτάξαμε την οικονομική αξία. Και μας είπαν οι εμπλεκόμενοι φορείς ότι το πλαστικό, η αξία του είναι μηδέν. Αυτό που έχει αξία είναι το ψηφιακό περιεχόμενο. Γι' αυτό είπαμε ότι θα ισχύσουν οι κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο, γιατί αυτό είναι το πραγματικό αντικείμενο που έχει αξία ε, όταν αγοράζεις ένα υλικό αγαθό με ψηφιακό περιεχόμενο. Γι' αυτό ε, πιστεύουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι που μπορεί να το κατανοήσει ο καταναλωτής. Αν πάω με το DVD μου στο κατάστημα δεν με νοιάζει αν υπάρχει κάποια ε, γρατζουνιά πάνω στο DVD. Εγώ αυτό που θέλω είναι να δω την ταινία. Άρα γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι θα ισχύουν οι κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και τέλος, ε, κυρία Γκέπχαρτ, αναφερθήκατε στην ε, τρισδιάστατη εκτύπωση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Που όμως ε, ασχολούμαστε εμεί με αυτό μόνο εν μέρη γιατί στο, στην τρισδιάστατη εκτύπωση ε, παίρνετε ένα ψηφιακό αρχείο και αν ε, συμβεί κάτι κακό ε, θα, ισχύσουν οι, οι κανόνες για, την ψηφιακού, για το ψηφιακό περιεχόμενο. Αν όμως το αντικείμενο που θα προκύψει από την τρισδιάστατη εκτύπωση, ε, τότε τα, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα ακόμα για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Είναι σημαντικό το θέμα, αλλά δεν θέλαμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα εδώ σε αυτή την πρόταση, γιατί απλά δεν έχουμε ακόμα επαρκείς γνώσεις. Και μετά ακούστηκαν και κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένες διατάξεις της πρότασης. Συγγνώμη, δεν κράτησα κάποια σειρά, απλά ε, απάντησα στις ερωτήσεις του, της κυρίας Φόρτ. Τι είναι, τι είναι αυτό το άλλα δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα είναι όρος σαφής. Γιατί ο, ο ορισμός υπάρχει στον σχετικό κανονισμό, όλα είναι, είναι σαφέστατα, οτιδήποτε μπορεί να ε, αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι προσωπικά δεδομένα. Any other data, άλλα δεδομένα είναι οτιδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε δεδομένο δηλαδή δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο, εμπίπτει σε αυτά τα άλλα δεδομένα και κατά συνέπεια σε αυτή την οδηγία. Ε, ερώτηση γιατί θα πρέπει να, να, η... η... να παρέχεται η υπηρεσία άμεσα. Η CRD λέει ότι θα πρέπει να παρέχεται το προϊόν ε, Εντό 30 ημερών. Αυτό όμω δεν έχει, δεν έχει νόημα για το ψηφιακό περιεχόμενο γιατί το ψηφιακό περιεχόμενο ε, παρέχεται άμεσα μέσω του, του ίντερνετ. Δεν χρειάζεται φορτηγό για να το μεταφέρει το ψηφιακό περιεχόμενο. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις όπου ο πάροχος μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα χρειαστεί χρόνο. Ε, στην ακρόαση ε, που είχαμε πριν, ακούστηκε το εξή. Αν ε, δεν έχει βγει ακόμα το καινούριο CD Αντέλ, αλλά εγώ έχω αγοράσει μια σύνδρομη, ο πάροχο γνωρίζει ότι δεν μπορεί ακόμα να παράσχει στους καταναλωτές το καινούριο CD τη Αντέλ γιατί δεν έχει βγει ακόμα αλλά θα μπορεί να το κάνει σε ένα μήνα γι' αυτό στην, ε, στο 5-2 λέμε εκτό αν τα συμβαλώμενα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά άρα δίνεται τη δυνατότητα στον πάροχο να λέει ότι εδώ θα πρέπει να σου παράσχω αυτή την υπηρεσία ή αυτό το, το αγαθό, το προϊόν ε, με κάποια καθυστέρηση. Και αυτό υπάρχει δυνατότητα στην οδηγία να, να το κάνει κανείς. Η ερώτηση του κυρίου Φως. Για το που υπάρχει ελευθερία ε, στη σύμβαση. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 19, όλες οι διατάξεις οδηγίας είναι κείμενο ε, δίκαιο και αναγκαστικό, δεσμευτικό. Δεν είναι στη διακριτική ευχαίρεια, ούτε μπορεί κανείς να το εφαρμόσει βάρος των καταναλωτών. Με δύο εξαιρέσεις. Μία αναφέρεται στο άρθρο 19 που υπάρχει η δυνατότητα αυτή, το άρθρο 5 παράγραφος 2 το είπα προηγουμένου και ε, ε, το άρθρο 6 ε, εδάφιο 4. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία εξαιρέσεων, είναι οι περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει διαπιστώσει το σφάλμα, ξέρει ότι είναι ελαττωματικό το περιεχόμενο το προϊόν, ξέρει και τα δικαιώματά του και πάει στον προμηθευτή. Τότε θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και οι δύο να συμφωνήσουν διαφορετικά αυτό υπήρχε και στην οδηγία την προηγούμενη για τα κατανολικά αγαθά και την έχουμε υιοθετήσει με το ίδιο σκεπτικό. Στη συνέχεια έγινε και μία ερώτηση, νομίζω από την κυρία Φόρτ, για πολύ ειδικού όρους που χρησιμοποιούμε στο άρθρο 6, παράγραφος 1, α, ε, λειτουργικότητα, διαλειτουργικότητα και ε, άλλα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να το αντιγράψουμε από τους κανόνες για το δίκαιο πολίσεων. Ε, συμφωνώ απολύτως και δεν το κάναμε. Αναφέρουμε συγκεκριμένα σημεία τα οποία βρήκαμε κοιτάζοντας και μελετώντας πολλές συμβάσεις και πολλά προβλήματα που έχουν οι καταναλωτές και είναι οι πιο συχνές κατηγορίες προβλημάτων. Διαλειτουργικότητα, λειτουργικότητα, ασφάλεια, προσβασιμότητα, συνέχεια Αυτά είναι οι διόψεις του ίδιου νομίσματος τα δύο τελευταία. Ουσιαστικά αυτά είναι τα βασικά προβλήματα και γι' αυτό το αναφέρουμε εκεί, ε, έχουν προβλήματα συχνά καταναλωτές με το ψηφιακό περιεχόμενο. Άλλη ερώτηση. Ο προμηθευτής θα πρέπει να επιστρέψει όλα τα δεδομένα στο πέρας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 30. Και αυτό με φέρνει σε διάφορες άλλες ερωτήσεις βουλευτών που έκαναν αντίστοιχα ερωτήματα, όπως η κυρία Κάλλας. Να σας εξηγήσω, αν θέλετε, πολύ σύντομα ε, το άρθρο 30. Στο B και στο C κάνουμε μία διάκριση μεταξύ εκείνων των δεδομένων που έχουν ε, πληρωθεί και ως αντίτιμο έχουν καταβληθεί για μια ε, άλλη υπηρεσία τους που, που τους παρέχεται. Και εδώ ο, ο προμηθευτής ε, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν προσωπικά δεδομένα και άλλου είδους δεδομένα. Έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να καλύψουμε και τα δύο. Λέμε λοιπόν στο άρθρο 30C ότι εάν ο προμηθευτής κάνει αυτό που κάνει για τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό CDPR, ε, δηλαδή ανωνυμοποίηση και τα λοιπά, είναι το ίδιο ε, που πρέπει να κάνει εδώ, δηλαδή να μην τα χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν όμως άλλα δεδομένα τα οποία έχει αγοράσει εντό αγωγικών ο προμηθευτής, γιατί είναι το αντίτιμο και δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί πια. Και μετά υπάρχει μια διάκριση στο C, που είναι το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο έχει παράσχει, για παράδειγμα έχω αποθηκεύσει στο cloud δεδομένα, φωτογραφίες για παράδειγμα, οικογενειακές. Μπορεί να είναι προσωπικά δεδομένα, συνδέεται αυτό με μένα ή με άλλο πρόσωπο της οικογένειάς μου, αλλά μπορεί να είναι και ένα γιοβασίλεμα ή ένα βουνό που έχω βγάλει φωτογραφία που δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Αναλύσαμε στο cloud computing ε, στην ομάδα πυρογνωμόνων πάρα πολλές συμβάσεις και βρήκαμε πολύ συχνά ρήτρες που επιτρέπουν στον προμηθευτή να τα χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό θέλει και πολλές φορές αυτό το λέμε πάρα πολλά λόγια. Δηλαδή μπορεί να κάνουν ας πούμε διαφήμιση με τη δική μου φωτογραφία του, του βουνού. Εγώ μπορεί να έχω συλλογή βασιλεμάτων ας πούμε ή νυχτερινές λήψεις ε, συγκεκριμένων ε, μνημείων ή ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Εάν ε, το έχω στο cloud και διαπιστώσω ένα ελάττωμα και θέλω να τερματίσω τη σύμβαση ε, και δεν έχω πρόσβαση σε αυτά, δεν μου επιτρέπει ο πάροχος να ασκήσω τα δικαιώματά μου. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να αποθαρρύνονται οι καταναλωτές ή να εμποδίζονται ε, να κάνουν χρήση των δικαιώματων τους επειδή δεν τους δίνουν πίσω το περιεχόμενο ή το, το δίνουν με τρόπο που να μην μπορούν να αλλάξουν πάροχο ή πρέπει να περιμένουν πολύ καιρό ή πρέπει και να πληρώσουν ακόμα. Αυτή είναι η λογική λοιπόν που κρύβεται από πίσω. Νομίζω έτσι απάντησα σε ορισμένα από τα σχόλια της κυρίας Κάλλας. Ρώτησε και κάτι άλλο η κυρία Κάλλας, τι γίνεται με τις πλατφόρμες που έχουν άλλα στοιχεία όπως είναι στοιχεία πληρωμών. Α, σταματώ εδώ διότι δεν θα προλάβουμε. Στο συγγνώμη. Μπορείτε να απαντήσετε την ερώτηση της κυρίας Κάλλας, αλλά πραγματικά έχουμε καθυστερήσει, δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Ζητώ συγγνώμη. Πλατφόρμες είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Ε, μπορεί να είναι πάροχος ή ενδιάμεσος. Ε, στην πρώτη περίπτωση καλύπτονται από την οδηγία αν όχι δεν καλύπτονται και επομένως δεν χρειάζεται να ε, συμμορφώνονται με τις απαιτήσει. Όμως επεξεργάζονται δεδομένα και ελέγχουν δεδομένα, οπότε υπό το GDPR ο καταναλωτής μπορεί να ε, κατηγορήσει την πλατφόρμα. Εγώ έκανα κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν απαντήθηκαν ο λόγος για τον οποίο έγιναν τόσο πολλέ ερωτήσει ήταν γιατί εδώ οι συνάδελφοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς, να, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Η Τζούλια που με ρώτησε για τα smartphones, ε, το αν καλύπτονται από την οδηγία ε, με, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ω υλικά αγαθά. Ίσως γραπτούς να μπορείτε να μας απαντήσετε σε κάποιες ε, ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα το θέμα των παρόχων, ε, ε, τηλεφορτωμένου περιεχομένου, ναι, βεβαίω. Μπορούμε να απαντήσουμε διμερό, λέει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, λέει η πρόεδρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις ε, πλατφόρμες Επιτροπής μας. Να δώσω τώρα το λόγο στο συνπρόεδρο. Μία ε, τελευταία ερώτηση προς τους συνεισηγητές. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ε, ποια είναι τα επόμενα στάδια και ένα χρονοδιάγραμμα ενδεχομένως. Η ε, κύριε Γκέφχαρτ. Ναι. Συναντηθήκαμε χθε με τον κύριο Φω, με τι γραμματείε των Διεπιτροπών και σα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μα. Στην αρχή είχαμε διαφορετική άποψη, αλλά τελικά τα βρήκαμε και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει ακόμα πριν το καλοκαίρι να έχουμε ένα έγγραφο εργασίας και βάσει αυτού τον Ιούλιο να κάνουμε μια συζήτηση και στις δύο επιτροπές κοινή για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η έκθεσή μας. Και για το Σεπτέμβριο να φέρουμε το σχέδιο έκθεσης και συγκεκριμένα 7 Σεπτεμβρίου θα τη δίναμε σε μετάφραση κανονικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες μας. Οπότε, από εκεί και πέρα προθεσμία για τις τροπολογίες, μάλλον να το πω αλλιώ. συζήτηση ε, για το σχέδιο 29 Σεπτεμβρίου, 13 Οκτωβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες και 7 και 8 Νοεμβρίου να συζητήσουμε τις τροπολογίες στις επιτροπές και διαπιστώσαμε ότι έχουμε διαφορετικές παραδόσεις η Γιούρη και η Ίμκο. Διότι στην ΙΜΚΟ, Επιτροπή Εσωτερική Αγορά, έχουμε πάει για τακτική να έχουμε και τι συμβαστικέ τροπολογίε που συζητούμε. Στη Γιούρι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα το χειριστούμε, γιατί έχουμε δει τι διαφορετικές παραδόσεις και ήθη και έθιμα. Υπάρχουν τώρα δύο δυνατότητε. Και δεν το αποφασίσω εγώ, πρέπει να το αποφασίσουν οι συντονιστές στην Επιτροπή Εσωτερικού και να μην το κάνουμε αυτό έτσι, αλλά αν ε, προηγουμένως συνεδριάσουμε ε, από κοινού με τους σκιώδεις συγητές. Εκτός της συνεδρίας δηλαδή της κανονικής το κάνουμε αυτό τακτικά. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο και στις 5 Δεκεμβρίου να ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης. Κάπως έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα. Σε αυτό συμφωνήσαμε, αν τα κατάλαβα καλά. Αλλά στο μεταξύ ο κύριος Φως έχει αλλάξει γνώμη και με εκπλήσει αυτό γιατί χτες νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει. Ελπίζω να ε, γίνεται να τα καταφέρουμε για να τελειώσει η εργασία μας στις επιτροπές εντός του έτους και το σύντομότερο να πάμε στην Ολομέλη αρχές του 17. Το αργότερο. Ο κύριος Φως. Πάρα πολύ σύντομα, συμπληρωματικά. Βεβαίως και συμφωνήσαμε ε, ε, σε περίπτωση που μας κατακλείσουν όμως τα προβλήματα ή με την άλλη πρόταση ή δεν τα βρούμε ή δεν συνεννοηθούμε και χρονικά, ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα να επιδείξουμε κάποια ευελιξία για να λύσουμε το πρόβλημα. Μια μικρή υποσημείωση είναι αυτή. Προς το παρόν το σχέδιο μας είναι ε, να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά αν δυσκολέψουν τα πράγματα μπορεί και να αλλάξει λίγο. Ευχαριστώ. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δίνω και πάλι το λόγο στον ε, κύριο Σφόμποντα. Κλείνουμε και το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης. Ο κύριος Σφόμποντα λέει ευχαριστώ Βίκη που συμπροεδρεύσαμε. Και περνάμε στο